το άρθρο 10 θέλαμε να το διαγράψουμε αν η συγχρηματοδότηση για τα κράτη-μέλη είναι πέραν των επιπρόσθων κονδυλίων θα είναι υπερβολικά επαχθή στη διαδικασία. Και εμείς είπαμε όχι, θέλουμε να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα για τα χρηματοδοτικά μέσα. Δεν θέλουμε να ε, υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στον προπολογισμό της Ένωσης και τη χρηματοδότηση των κρατών μελών. Γι' αυτό προτείνουμε διαγραφή του άρθρου 10. Υπάρχουν και άλλες ε, προτάσεις και θα μας βοηθούσε να μας πείτε πώς ακριβώς θέλετε να κινηθούμε στο μέλλον να μας βοηθούσε για τις μελλοντικές συζήτησεις κατά τη γνώμη μου. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πολλές τροπολογίες κινούνται προς την κατεύθυνση να συμπεριληφθούν διοικητικές αρχές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Έχουμε κάνει υποβάλει ήδη μια τροπολογία σε σχέση με τον ορισμό εξ αρχής και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές ε, ε, συμπεριλαμβάνονται. Δεν χρειάζεται λοιπόν να μπλέκουμε γραφειοκρατικά, με απλές κινήσεις μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε αυτά από πλευράς μου και το ταχύτερο δυνατόν θα οργανώσουμε τις, ε, τις συνεδρίες των σκιωδών για να συζητήσουμε τις συμβαστικές. Αλλά θα, πραγματικά θα ήθελα να ακούσω τη σχόλια από την Επιτροπή για το άρθρο 10. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήδη μάλλον αποκαταστάθηκε και η διερμηνία, τα κανάλια που είχαν κάποιο πρόβλημα. Ο κύριος Βανίστελ θα ήθελε. Ε, κοιτάξτε, η συνάδελφος ανέφερε ακριβώς τα σημαντικά θέματα. Και η δική μας προσέγγιση για όλες αυτές τις τροπολογίες δεν αφήνει κάποια ερωτηματικά επί του μέσου μόνο λεπτομέρειε, δηλαδή τα, σημαντικά τα ανέφερε ήδη Κωνσταντ. Τώρα, η, η Κομισιόν πρέπει να προχωρήσει ταχαίω. Αλλά ήθελα το εξή να θίξω. Μετά την ψηφοφορία του Νοεμβρίου, θα μπορούσαμε να έχουμε μια εντολή διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο ώστε να γίνει αυτό για να μην πρέπει να παραπέμπουμε κάθε φορά στην Ολομέλεια ούτω ώστε τον Απρίλιο να έχουμε αποτελέσματα και ούτω καθεξής. Το λέω γιατί όπως ξέρετε και άλλες επιτροπές είχαν απορίες σχετικά με τον ηγετικό ρόλο της ΡΕΓΚΙ και εμείς καθυστερήσαμε και καλό θα ήταν να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Οπότε το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι δεν θέλουμε να χαθεί άλλος χρόνος. Γιατί ίσως μπορεί να ληφθούν υπόψη κάποιες καλές ιδέες. Δηλαδή είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό. Μάλιστα και ο Βανίστελόι. ο κύριος Νοβάκοφ ε, μετά η κυρία Ρένκε α, θέλετε να φύγετε ο κύριος Γιάφκητσης ε, ο οποίος ε, θα, θα χρειαστεί να φύγει μετά α, στο ίδιο μέρος θα πάτε μάλιστα η κυρία Τόμασιτς και μετά ο κύριος Γιάκοφτσης Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι πρέπει να πάω στην συνάντηση της ΠΕΣΟ και καθότι είμαι σκιώδης ήθελα να πω τα εξής. Οι διαθετικές μεταρρυθμίσεις σε οποιαδήποτε περιοχή πολιτικής είναι πολύ σημαντική πρόκληση γιατί χρειάζεται χρόνος για να δει κανείς τα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου είναι κρίσιμης λεπτομέρεια, ε, με συγχωρείτε, να έχουμε αταχαίω αποτελέσματα. Και για να ε, έχουμε αποτελέσματα από το άρθρο 4, χρειαζόμαστε τη, τη συνεισφορά των δημοσίων φορέων ώστε να ληφθούν υπόψη μάλλον ώστε να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα και ώστε να υπάρχουν και οι κατάλληλες αρμοδιότητες για την υλοποίηση των πολιτικών μεταρρυθμίσεων και για την καλύτερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. Στις τροπολογίες μας λοιπόν και εγώ στη δική μου ήθελα αυτό ακριβώς να βελτιώσω την ε, διοικητική και διαχειριστική ικανότητα των τοπικών και περιφερειακών φορέων και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να συμπεριλάβουμε όλα τα επίπεδα διοίκησης η στήριξη των τοπικών και περιφερειακών φορέων είναι πολύ σημαντική ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και οι επενδύσεις ε, συνολικά στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης συμπεριλαμβανομένης και της ε, βοήθειας για την αποτελεσματική χρήση των ε, ενωσιακών πόρων. Ήθελα επίσης να τονίσω το θέμα της διαφάνειας και της καλή διακυβέρνηση είναι εξαιρετικά σημαντικό ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των δικαιούχων άλλων κρατών μελών και της Κομισιόν. Αυτή η αμοιβή εμπιστοσύνη όμως δεν μπορεί να ενισχυθεί εφόσον δεν υλοποιήσουμε αποτελεσματικά τις μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Μάλιστα. Ο κύριος Γιάκοφτσιτς τώρα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί έχω και εγώ αντίστοιχη υποχρέωση και δεν θα μπορέσω να συμμετάσχω περισσότερο. Ε, ήθελα να πω ότι λυπούμεθα που διαγράφει η πρόταση Κομισιόν. Εμείς υποβάλαμε την τροπολογία μας ώστε να επανέλθει το τμήμα που διαγράφει από την πρόταση Κομισιόν. Θεωρούμε λοιπόν ότι η τεχνική βοήθεια που θα μπορούσε να είναι υποφελής για τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα, να επανέλθει μάλλον. Γιατί κατά τον τρόπο αυτόν θα μπορούσαμε να επιτύχουμε κάποιες ε, συνέργειες. Θα έλεγα λοιπόν ότι καλό θα ήταν να γίνουν αποδεκτές οι τροπολογίες μας και να επανέλθει η αρχική πρόταση. Δεν θέλουμε τροπολογίες που διαγράφουν τα πάντα. Αυτό ήθελα κυρίως να τονίσω. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Ρένκε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους ε, συνεισηγητές αλλά και τους άλλους συναδελφούς. Πολύ σύντομα να επανέλθω στην συζήτηση που είχαμε από την αρχή που είναι πολύ σημαντικό. Μετά την αποστολή στην Ελλάδα με την αντιπροσωπεία της ε, Ρέγκη εγώ επιβεβαιώθηκα στο εξής πρέπει να αποφύγουμε ότι αυτό φαίνεται σαν να υποσκάπτουμε αργά αλλά σταθερά την πολιτική συνοχή. Εμείς ως Επιτροπή Ρέγγι πρέπει να καταστήσουμε σαφέστατο με το σχέδιο έκθεσής μας και με την έκθεση που τελικώ θα εγκριθεί ότι έχουμε εμπιστοσύνη ότι η πολιτική συνοχή με τις αρχές της πολιτικής αυτής, με τους εταίρους, με τις ε, συνεργατικές μορφές της ε, Κοινωνία των πολιτών με το όλο πρότυπο διαχείρισης δεν επιβάλλει άλλο άχθος στις περιφερειακές ε, αρχές αλλά τις ενισχύει και τις βοηθάει. Αυτό είναι η κρίσιμη σημασία αν είναι να λειτουργήσει στο τέλος. Οι ελληνικές τοπικές αρχές μας κατέστησαν σαφέστατο ότι προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αυτό είναι καλό, χρήσιμο εργαλείο. Αλλά δεν πρέπει να επιβληθούν άλλα σκεπτικά σχετικά με μεταρρυθμιστικές τροποποιήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθούν. Και με την ε, μακροαιρεσιμότητα το ίδιο είχαμε συμφωνήσει. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό θα μπορούσε πράγματι να διευκολύνει τις τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς όχι ως εργαλείο τιμωρίας, αλλά ως μέσο διευκόλυνσης. Πρέπει λοιπόν να επιτύχουμε μια ισορροπία και περιμένουμε ενδιαφέρον τις περαιτέρω συζητήσεις που θα έχουμε. Πρέπει να επιτύχουμε πάντως μια σωστή και ξεκάθαρη ισορροπία και το ίχνος της Επιτροπής μας πρέπει να είναι σαφέστατο στην όλη αυτή η τροπολογία ώστε να παραχθεί η βοήθεια αυτή στα κρατημέλη και από εκεί και πέρα με μεγάλη χαρά να το υποστηρίξουμε όσο άλλο μπορούμε. Αλλά θα πρέπει να, ε, όπως έχουν υποβληθεί, να γίνουν διάφορες προτάσεις ε, στο σχέδιο για να δουλέψουμε επικοδομητικά. Μάλιστα, σε ευχαριστώ. Κυρία Μάτο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξετάζουμε τις τροπολογίες ε, μια προτάσεως τη Επιτροπής και ήθελα να σα εξηγήσω γιατί εγώ και η αντιπροσωπεία μου προτείναμε την διαγραφή της προτάσεω. Πρόταση που υποβάλλεται για τις μεταρρυθμιστικές για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. 140 τόσα εκατομμύρια ευρώ για τις μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα υπό το άρθρο 5 και υπογραμμίζω ποιες είναι, εκπαίδευση, κατάρταση, απασχόληση, κοινωνική συμπερίληψη, κοινωνική αρρωγή και βοήθεια, ε, δημόσια υγεία, όλα αυτά μας φαίνονται απολύτως αντίθετα στις βασικές αρχές της ε, εδαφικής ε, συνεργασίας και της πολιτικής κοινωνικής συνοχής. Στην περίοδο 14-20 με τη θεματική 11 έχουμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ που θα γίνουν 6,5 με την εθνική συμμετοχή. Επομένως, γιατί υποβάλλει την πρόταση αυτή. Τι βρίσκεται από πίσω, ποια είναι η πολιτική ατζέντα που κρύβεται πίσω από αυτό. Εμείς με, ε, ε, επί της εκθέσεως της κυρίας ε, Τόμασιτς θα συζητήσουμε τι δεν λειτουργεί τεχνικά. Ξέρετε ότι εγώ πάντοτε επέκρινα τα προβλήματα που έχουμε στη δική μας ε, χώρα, τονίζοντας συνεχώς ότι χρειαζόμαστε αναβάθμιση και στην απορρόφηση των κονδυλίων, αλλά και στην ποιότητα των δαπανών. Όμως, στην πρόταση αυτή πηγαίνουμε πολύ πέραν αυτού. Οι συνάδελφοι εισηγητές έχουν προβεί σε μία, μάλλον, εγώ έχω εξετάσει τις τροπολογίες που υπέβαλαν συνάδελφοι, η τροπολογία 40 παραδείγματι θα ήθελε να διαγραφεί η παράγραφος 10 της προτάσεως, ώστε να χρηματοδοτείται το πρόγραμμα μέσω συνεισφορών επιπρόσθετων από εκείνες των κρατών μελών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι και οι ίδιοι εκφράζουν την ανησυχία το πρόγραμμα αυτό να γίνει κάτι σαν πασπαρτού για τις ε, ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όπως και άλλες ε, τροπολογίες, όπως η 20 αν ακούσαμε καλά, για την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος εκπαίδευση, ή εκείνη τη κυρία Ρένκε που προτείνει να είναι τα κράτη-μέλη που θα καθορίζουν από κοινού με τις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές. Αυτές οι τροπολογίες όμως δεν υπαρκούν, διότι ο λόγος, το κλάσμα μας ανησυχεί ιδιαίτερω. Στην ίδια τη φύση της προτάσεω και με τα λόγια του Αντιπροέδρου Ντονκόφσκι υπάρχει μια απόπειρα τιμωρία και άλλη εμπασχευτός κατεύθυνση για διάφορα κράτη-μέλη και χρηματοδότηση ε, μεταρρυθμίσεων που στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Γαλλία έχουμε μαζικότατες διαδηλώσεις. Θα είναι ένα πολύ κακό σημάδι, μήνυμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους πολίτες της. Δηλαδή είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα για μια καταστροφική μεταρρύθμιση μετά το 2020 και επιφυλασσόμενοι ε, για την αξία κάποιων συγκεκριμένων τροπολογιών εμείς προτείνουμε την απόλυτη απόσυρσή τους. Ε, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Νοβάκοφ δυστυχώς έφυγε από την συνεδρίαση γιατί είχε άλλα, άλλες δεσμεύσεις. Ε, κύριε Μπότσακ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Δεν θέλω σε σχέση με αυτή την πολιτική ή και σε σχέση και με την χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος σε σχέση με τις διαθροτικές μεταρρυθμίσεις που προέρχονται αυτές ε, οι δράσεις από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη δυνατή λύση. Όμως για το μέλλον θα πρέπει να εξετάσουμε <clears throat> το πρόγραμμα αυτό να είναι ανεξάρτητο στη χρηματοδότησή του ώστε σε σχέση με την ε, πολιτική συνοχή, σε σχέση με τη δομή του να ε, μπορεί να έχει τη σωστή θέση. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για τις ε, τροπολογίες και γι' αυτό αισθάνομαι την υποχρέωση συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να αναφέρω την πρόταση για την διαθροτική μεταρρύθμιση στοχεύει στο να διασφαλιστεί η δυνατότητα των διαθετικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο ακόμα και εκείνων των ε, μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται από τις προϋποθέσεις και όρους ε, για τον μηχανισμό χρηματοδότησης. Είναι σημαντικό ότι οι εξάντε εκ των προτέρων ε, προϋποθέσεις και όροι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ακούσαμε και από πλευράς Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι τόσο χαμηλή η απορρόφηση σε σχέση με την διάθεση των διαθωτικών προγραμμάτων είναι επειδή υπάρχουν αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις και η δυνατότητα των κρατών να ε, αντιδράσουν και να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτούς όλους και προϋποθέσεις είναι περιορισμένη. Θα πρέπει λοιπόν εδώ το θέμα αυτό να ληφθεί υπόψη σε σχέση με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών. Πρέπει να υπογραμμίσουμε αυτή την πτυχή. Γι' αυτό κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στην Ελλάδα, στην Αθήνα, είδαμε τα θετικά αποτελέσματα τέτοιου είδους προγραμμάτων σε αυτό το συγκεκριμένο κράτος μέλος ε, στην ε, Ελλάδα και σε σχέση με το, το πώς λειτουργούν εκεί τα πράγματα το είδαμε σε σχέση με την ε, επίσκεψή μας εκεί. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα λοιπόν να υλοποιήσουν τα αναγκαία μέτρα για την ανταποκρίνονται στους όρους και προϋποθέσεις όπως και σε αυτό το πρόγραμμα και, ε, στο πρόγραμμα συνοχής ε, ε, και όσον αφορά την χρήση της τεχνικής αρρωγής όσον αφορά τα εν λειτουργία προγράμματα Υποστηρίζω την κυρία Κράιλ προς την ερώτη... για την ερώτησή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το είδαμε αυτό, είναι χρήσιμο. Το είδαμε στην Ελλάδα ήδη. Δεν βλέπουμε να υπάρχει κάτι πίσω από αυτό το μέτρο. Υπάρχει απλώς η επιθυμία να υποστηριχθούν οι μεταρρυθμίσεις και να μπορέσουν αυτές να προαχθούν ώστε τα κράτη-μέλη να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν με καλύτερο τρόπο τα κονδύλια των διαθροτικών ταμείων. Θα πρέπει όμως να έχουμε περισσότερες επεξηγήσεις και να δοθούν παραδείγματα σχετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το χαιρετίζαμε ιδιαίτερα ως ευκαιρία για τα κράτη-μέλη, παρότι θα ήθελα να υπογραμμίσω εδώ και πάλι ότι είναι απόλυτα μια θετική εμπειρία αυτή που ε, βιώσαμε και είδαμε. Και δεύτερον, είναι θέμα ε, της ε, επιθυμίας να υπάρξει ανταπόκριση από πλευρά συγκεκριμένου κράτους μέλους. Αυτά ήθελα να πω και εκτιμώ την ε, εξέλιξη αυτού του διαλόγου και ελπίζω ότι από πλευράς εισηγητών θα υπάρξει ανοιχτό πνεύμα για κάποιες προτάσεις ε, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε. Αυτά ήταν όσα είχα να πω. Και τώρα για να, να δώσουμε τον λόγο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε την κυρία Μακάρθη. Έχετε τον λόγο παρακαλώ λοιπόν. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να επεξηγήσω περαιτέρω το θέμα για την χρηματοδότηση και το άρθρο 25. Ζητώ συγγνώμη για τις παρεμηνίες ε, και παρεξηγήσεις. Επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να επεξηγήσω το θέμα αυτό. Φυσικά έχετε ε, γνωρίσει την, τις προκαταβολές ως δυνατότητα δράσης. Είναι ένας τρόπος που τα κράτη-μέλη μπορούν να έχουν την επιλογή σε σχέση με την συγχρηματοδότηση από πλευράς τους. Όμως στη δική μας πρόταση δεν υπάρχει επιλογή για τα κράτη-μέλη μέσα σε αυτό το πλαίσιο για τη συγχρηματοδότηση. Και γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό συμβαίνει διότι τα χρήματα τα οποία διαθέτουμε για την τεχνική αρρωγή δεν τα παρέχουμε στα κράτη-μέλη. Τα κονδύλια αυτά <clears throat> διατίθενται στους ε, παρέχοντες αυτές τις υπηρεσίες. Δεν υπάρχουν λοιπόν παρόμοιες ευκαιρίες για τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν σε αυτό το πλαίσιο από πλευράς τους ο τρόπος με τον οποίο εσείς εννοείτε την συγχρηματοδότηση δεν είναι μέρος αυτού του προγράμματος. Δεν πάνε τα χρήματα άμεσα στα κράτη-μέλη, πάνε στους παρόχους που παρέχουν αυτή την τεχνική αρρωγή. Τώρα για να μπορέσουμε να το αποφύγουμε, να το παρακάμψουμε αυτό, να το υπερβούμε, σε σχέση για παράδειγμα και με την Ελλάδα και την Κύπρο υπήρξε μια τροπολογία ε, η οποία αναφερόταν στο άρθρο 25 και αυτή η τροπολογία, με αυτή την τροπολογια κάτι κράτη-μέλη που βρίσκονται υπό ένα πρόγραμμα προσαρμογών οικονομικό από την δική τους, ε, μέσω δικής τους επιλογής, όχι υποχρεούμε, δεν υποχρεούνται, θα μπορούν να μεταφέρουν κονδύλια από την αρρωγή ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται εξ ονόματός τους ε, για λογαριασμό τους, ε, για προγράμματα τεχνικής αρρωγής στα οποία έχουν συμφωνήσει. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο υποχρεωτικό πλαίσιο, κάποια περιστολή, κάποια, κάποιος καταναγκασμός. Ε. <clears throat> Δεν ζητάμε από τα κράτη-μέλη, δεν επιβάλλουμε να διατεθούν αυτά τα χρήματα σε σχέση με την τεχνική αρρωγή. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα στην περίπτωση της Ελλάδας, το 2014 επιστρέψαμε 50 εκατομμύρια ώστε να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με τις ελληνικές αρχές ώστε να μπορέσουν οι ελληνικές αρχές ε, να ε, συνάψουν συμβόλαια και να πληρώσουν παρόχους τεχνικής αρρωγής. Μας επέστρεψαν οι ε, ελληνικές αρχές 13 εκατομμύρια για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι όροι και προϋποθέσεις ως ορόσημα που έπρεπε να επιτευχθούν για να ανταποκριθούν οι Έλληνες σε αυτό το πρόγραμμα. Αντίστοιχα στην Κύπρο. Ποια είναι η πρόθεσή μας λοιπόν σε αυτή την πρόταση. Η πρόθεσή μας είναι να προσφέρουμε αυτή την επιλογή και σε άλλα κράτη-μέλη. Είναι μια επιλογή, δεν, είναι, δεν επιβάλλουμε αυτή την επιλογή είναι μια επιλογή που είναι ελεύθερη στα κράτη-μέλη αν αποφασίσουν να επιστρέψουν κάποια κονδύλια και αυτά τα κονδύλια τα οποία θα επιστρέφονται θα βρίσκονται υπό τον απόλυτο έλεγχο των εμπλεκομένων κρατών μελών ώστε η τεχνική αρρωγή η οποία έχει με συμβόλαια, με συμβάσεις συναυθεί να είναι κάτι επί του οποίου συμφωνούν αυτά τα κράτη-μέλη. Δεν είναι κάτι λοιπόν το οποίο επιβάλλουμε. Επιτρέπει συνέργειες αυτή η δυνατότητα γιατί. Διότι, για παράδειγμα, εφέτος κατά τη διάρκεια των προκατακτικών δράσεων έχουμε 3 εκατομμύρια. Τώρα τα 3 εκατομμύρια δεν είναι πολλά σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Είναι μια πρόταση για να βελτιωθούν τα πράγματα. Ωστόσο σε μεγάλα σχέδια τα χρήματα αυτά πράγματι θα είναι χρήσιμα θα μπορεί να είναι χρήσιμη αυτή η δυνατότητα. Αν δουν τα κράτη-μέλη ότι έχουν τη δυνατότητα έτσι να δράσουν, θα είναι υποφελές ε, για, αυτά... για αυτά τα κράτη να πούν «Ακούστε, δεν θέλουμε να περάσουμε όλες αυτές τις διεργασίες για να συναυθούν συμβάσεις για την τεχνική αρρωγή. Θα σας δώσουμε εσάς αυτά τα χρήματα και εσείς με σύμφωνη δική μας γνώμη θα προχωρήσετε σε αυτές τις ρυθμίσεις και διευθετήσεις είναι μια δυνατότητα που μπορεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να προσθέσουν κονδύλια στα δικά μας με αυτά τα οποία διαθέτουμε εμείς ώστε να μπορέσει να διατεθεί η τεχνική αρρωγή εκείνη που επιθυμούν τα ίδια αυτά τα κράτη-μέλη να τους χορηγηθεί. Θέλω να το τονίσω αυτό σε σχέση με αυτή την πρόταση. Δεν υπάρχει καθόλου υποχρεωτικός χαρακτήρας σε αυτή την πρόταση. Εμείς μπορούμε να δράσουμε μόνο όταν θα έχει διατυπωθεί το αίτημα από ένα κράτος μέλος. Δουλειά λοιπόν είναι του κράτους μέλους ε, να διατυπώσει ένα τέτοιο αίτημα, αν επιθυμεί αυτό να την χάνει της τεχνικής αυτής αρρωγής ε, <clears throat> δεν κρύβεται κάτι πίσω από αυτή την πρόταση ώστε εμείς να ε, το κάνουμε αυτό. Η βούληση και η πρόθεση θα είναι του κράτους μέλους και η επιλογή δική του. <clears throat> Γι' αυτό θα θέλαμε πραγματικά αυτή, αυτό το ειδικό άρθρο να διατυπώνεται και να εντάσσεται με αυτόν τον τρόπο, διότι δεν βλάπτει. Είναι μια ελεύθερη επιλογή. Δεν είναι κάτι το οποίο επιβάλλουμε εμείς υποχρεωτικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, υπάρχουν κάποια σχόλια ή είσαστε ικανοποιημένοι. Ναι, κύριε Φανίστερ Ρόι, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν δεν θέλουν συνάδελφοι να παρέμβουν, επιτρέψτε μου με βάση τα στοιχεία πληροφόρησης που μας δόθηκαν να πω ότι η διαγραφή του άρθρου 10 ήταν εκείνη που είχε ως σκοπό να περιορίσει το νέο μέσο στους στόχους που ετέθησαν και σε σχέση με τις πληροφορίες για το άρθρο 12 Ίσως υπήρξε μια παρανόηση, αλλά στο άρθρο 12 η συγχρηματοδότηση θα μπορεί να είναι μέχρι 100% των, του αρχικού κόστους χωρίς αυτό να, ε, ε να συμμορφώνεται σε κάποιους όρους και προϋποθέσεις. Έτσι λοιπόν υπάρχει δυνατότητα αν κάποιο κράτος μέλος επιθυμεί να κάνει κάτι περισσότερο μπορεί να επιλέξει το ποσοστό εκείνο, ας πούμε το 20% και να το πληρώσει στους παρόχους τεχνικής αρρωγής. Ε, εδώ έγινε το αντίστροφο. Δεν ήταν αυτό κάποια ταχυδακτηλουργική ε, παρέμβαση. Είναι μια ομαλή διαδικασία ως ήθιστε και θα πρέπει αυτό και στις, ε, σε σχέση με την επεξήγηση που δόθηκε να αναφερθεί ότι πράγματι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση σε σχέση με αυτή την ε, δράση. Πρόκειται για τα πόσα χρήματα διατίθενται στο νέο αυτό μέσο. Αυτό είναι η μία φάση. Η άλλη πλευρά είναι πώς αυτά τα χρήματα θα μπορέσουν να διατεθούν, υπό ποιε προϋποθέσεις. Θα μπορούν να είναι 100% ή 80% αλλά εδώ υπάρχει ε, συμφυρμός και των δύο αυτών κειμένων στην ίδια σελίδα. Θα πρέπει να ε, στοχαστούμε να δούμε τι θα πρέπει να γίνει μελλοντικά. Αν εσείς το λέτε με τέτοια σαφήνεια ότι είναι εθελοντικού χαρακτήρα αυτή η δράση. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία θα διατεθούν για τη νέα περίοδο 2014-2020 για αυτή τη δημοσιονομική περίοδο με χαρά θα ε, διαπιστωθεί ότι θα υπάρχει μεγαλύτερο πλαίσιο για αυτή την τεχνική αγορά Τώρα όταν αυτά τα νέα κονδύλια θα περάσουν στο νέο μέσο, λέτε μάλιστα μπορούμε να διαθέσουμε και περισσότερα, να κάνουμε και περισσότερα. Και εδώ αφορά αυτό ένα από τα μελήματα της ομάδας μας Ίσια, για την εταιρική σχέση, διότι τα χρήματα τα οποία εγγράφονται σε αυτή τη δράση δεν ε, υπάρχει σε σχέση με την εξέβρεση συνένεσης μια μαγική λύση ή συνταγή εδώ λοιπόν θίγεται ένα κέριο σημείο του δεοντολογικού κώδικα του τρόπου δηλαδή με τον οποίο πρέπει να εργάζεται κανείς με την αποκεντρωμένη ε, με τον αποκεντρωμένο φορέα ή οργανισμό. Πρέπει να δούμε εδώ λοιπόν πόσο ισχυρή θα είναι η διατύπωση του ενός ή του άλλου και μπορεί να εξευρεθεί ίσως ένας συμβιβασμός. Εσείς ε, το βλέπετε έτσι, αλλά δεν πρέπει να είναι το τέλος αυτό. Όταν ε, δίνονται χρήματα για την, ε, τις δράσεις αυτές και, το, και πούν οι περιφέρειες ότι όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό, διότι τα χρειαζόμαστε αυτά τα κονδύλια για τους στόχους που πρέπει εμείς να υλοποιήσουμε. Αυτό είναι εκείνο το οποίο θα ήθελα με τους σκιώδεις εισηγητές να εξετάσουμε, να συνεξετάσουμε, να δούμε αν μπορεί να εξευρεθεί ένας ε, συμβιβασμός. Δεν είναι θέμα αρχής, αλλά είναι θέμα κατανόησης και ερμηνείας. Είμαι βέβαια ότι μπορείτε να βρείτε μια λύση μεταξύ των σκιωδών εισηγητών και των συνεισηγητών, διότι αυτό δεν είναι θέμα ουσίας ή πολιτικής ή αρχής, ε, είναι θέμα διαφορετικών ε, οργανισμών, ιδιαίτερα εδώ σε σχέση με τις ε, περιφερειακές και τοπικές αρχές και ε, το πώς θα διοργανωθούν αυτά σε σχέση με τους φορείς των κρατών μελών από ό,τι κατανόησα η τελευταία σας ερώτηση είναι πώς θα μπορέσει να συμβαδίσει, να ευθυγραμμιστεί η επιθυμία των τοπικών αρχών να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα για την τεχνική αρρωγή και από την άλλη να συγκεράσουμε την επιθυμία της κεντρικής εξουσίας για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι ένα θέμα των κρατών μελών. Δεν πιστεύω ότι είναι θέμα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί εκείνη να επιλέξει το ένα ή το άλλο ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν και να ευθυγραμμιστούν τα κράτη-μέλη. Ίσως, ίσως μπορεί να γίνει και αυτό, δεν το, δεν το γνωρίζω, δεν είμαι βέβαια, αλλά πιστεύω ότι μέσω των συζητήσεων των σκιωδών εισηγητών και συνεισηγητών θα μπορέσει να εξευρεθεί μια λύση και χαίρομαι που σήμερα μας δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες. Θέλετε να αντιδράσετε, να τοποθετηθείτε σαν όσα είπε ο κύριος Φανίστερ Ρόι. Ναι, για μας είναι θέμα επικουρικότητας ε, των κρατών μελών. Και αυτά είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε. Είναι ε, η διαδικασία λήψη αποφάσεων κάθε κράτους μέλους. Θέλω όμως να τονίσω πως όταν ασχολούμαστε με την παροχή τεχνικής αρρωγής. Συνεργαζόμαστε με όλα τα επίπεδα, περιφερειακό και τοπικό συμπεριλαμβανομένου. Όταν λοιπόν χρειαζόμαστε, ε, υπάρχει ανάγκη για τεχνική αρρωγή και προσπαθούμε να την παράσχουμε, συζητούμε με το πιο ενδεδειγμένο επίπεδο, τοπικό ή περιφερειακό, ανάλογα με τις ανάγκες. Τα κράτη-μέλη όμως παίρνουν τις αποφάσεις για τη βοήθεια από τα διαστατικά ταμεία ανάλογα με την ε, οικία οργάνωση. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Ευχαριστούμε. Θα... Ε, ο Βανίστερα. Κυρία Ρέτκη, εσείς ε, ξεκάθαρα απορρίψατε τη θέση δεν υπάρχει δυνατότητα συμβιβασμού. Εσείς είπατε πως είναι ευρύτερο αυτό το εργαλείο σε σχέση με την πολιτική. Εμείς συμφωνήσαμε να είναι ευρύτερη η χρήση αυτού του μέσου, διότι υπάρχει πλέον υπέρβαση του συνολικού στόχου. Ανάπτυξη θέση εργασίας και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με στην έκθεση του άρθρου 63, τα τρία βλέπουμε τα τρία τέταρτα των, ε, αναχώρα, ε, των ειδικών αναχώρα συστάσεων σχετίζονται με τη, τα θέματα πολιτικής συνοχής. Και κάποια άλλα με τις τράπεζες, τραπεζικό σύστημα. Οπότε ναι, ναι, ναι, είναι ευρύτερο το μέσο αυτό και γι' αυτό ασχολείται διαφορετική υπηρεσία με αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζουμε όμως να μπορέσετε να μας βοηθήσετε για να βρούμε ε, μια συμβαστική λύση, γιατί πώς θα γεφυρώσουμε το χάσμα. Ε, συγγνώμη Πρόεδρε, γιατί μου απίφθινε αυτό το σχόλιο άμεσα ε, και πρέπει να απαντήσω. Μα τι, έχουμε εδώ σύσκεψη σχεδόν. Δεν είμαι σίγουρη ότι πρέπει να το δεχτώ. Τέλος πάντων, τέλος πάντων, επειδή σας απίφθηνε άμεσα το λόγο, παρακαλώ στις τροπολογίες μας κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις πώς θέλουμε να οριοθετήσουμε τη χρήση και για τις ειδικέ αναχώρες συστάσεις προτείνουμε να είναι οι κατάλληλες συστάσεις ε, για κάθε χώρα και αυτή ήταν η πάγια θέση της Ρέτζη. Προσοχή, δεν θέλω εγώ να υπονοήσω πως κάποιος εδώ μέσα έχει κρυφές προθέσεις. Στην κρίση όμως διαπιστώσαμε ότι ε, δεν ήταν ξεκάθαρη η αιτιολόγηση κάποιων πολιτικών αποφάσεων και γι' αυτό επιδιώκουμε να είναι εποφελής ε, η διαδικασία για όλους, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το Κοινοβούλιο, για τα κράτη-μέλη. Πώς, πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί, πώς ε, θα επιτύχουμε χρηστή διαχείριση των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων ε, ζητώ συγγνώμη αν είμαστε καχύποπτοι, ζητώ συγγνώμη και αν δεν ακολουθούμε τη τη προταθή σε γραμμή, αλλά δεν είναι και αυτό μέρος του δημοκρατικού διαλόγου. Προτού αποφασίσουμε ποια ρότα θα ακολουθήσουμε, παρόλα αυτά εγώ παραμένω αισιόδοξη. Θα καταλήξουμε πιστεύω σε συμβαστικές λύσεις μετά το διάλογο. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Τώρα ε, έχουμε μια σαφή εικόνα σε σχέση με το τι μέλη γενέστε στη συνεδρία των ε, σκιωδών. Ε, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η θέση των φιλελευθέρων. Δεν είναι όμως ε, εδώ ο σκιώδης μας, οπότε έπρεπε να το αναφέρω και αυτό. Λοιπόν, πέρασε συζήτηση. Ελπίζω να βρεθούν συμβαστικές λύσεις. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Παρουσίαση Μία μελέτη του Policy Department B για τα προσαρμοσμένα προγράμματα εδαφική συνεργασίας από το Κέντρο Τεκμηρίου του Κοινοβουλίου δηλαδή. Έχουμε δύο συναδέλφου που θα μα παρουσιάσουν τη μελέτη, ο Νίκο Βαμπριάνη και ο Φρανσό Λιβέρ, Νίκο Φρανσό Λιβέρ. Θα σας δώσω το λόγο. Θέλω μόνο να επενθυμίσω στα μέλη της Ρέτζη πως εμείς τη ζητήσαμε αυτή τη μελέτη. Έχουμε εμπειρία ε, σε σχέση με την ε, έγκριση έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας ε, για την εδαφική συνεργασία και γι' αυτό θέλουμε να δούμε ακριβώς πώς λειτουργεί στην πράξη η εδαφική συνεργασία. Κύριε, έχετε το λόγο. Νίκολα Βουριάννη λέγομαι και ο, ο Φρανσουά θα με βοηθήσει για να σας παρουσιάσουμε τα απορίσματα αυτής της έκθεσης. Θα... Ποιος είναι ο γενικότερο στόχο, ποια είναι η μεθοδολογία και μετά ε, θα μπούμε στα, στις λεπτομέρειες, στα ευρήματα, ε, πορίσματα και συστάσεις της έκθεσης. Πρώτα απ' όλα. Ε, τα στοιχεία που χρησιμοποίησαμε Εδαφική συνεργασία είναι ένας από τους δύο στόχους της πολιτικής συνοχής. 10 δις ευρώ, 2,5% του συνολικού προπολογισμού της πολιτικής συνοχής για χρηματοδότηση πάνω από 100 προγραμμάτων. Ο γενικότερος στόχος είναι να χρηματοδοτηθούν κοινέ δράσει με βλεκόμενου φορείς από διάφορες χώρες. Ποιο, ποιος ο στόχος αυτής της μελέτης? Να αξιολογήσουμε κάποια από τα νέα στοιχεία του κανονισμού, του κανονισμού δηλαδή ETC για την εδαφική συνεργασία και πώς εφαρμόστηκαν στα συγκεκριμένα προγράμματα. Ιδιαίτερη έμφαση προσδώσαμε στην αξιολόγηση της ικανότητας των προγραμμάτων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις εδαφικής συγκέντρωσης και να προσδιορίσουν, να εντοπίσουν σε πιθανές συνέργειες με άλλα εργαλεία. Αναλύσαμε την ε, ικανότητα και τη χρήση από πλευράς των προγραμμάτων ε, καινοτόμων εργαλείων. Θα δούμε συνέχεια ποια εννοώ. Επίσης, ε, προαιρετικές ρυθμίσεις ε, του κανονισμού για να απλοποιήσουν τη διαδικασία για τα προγράμματα και για τους δικαιούχους. Ποια μεθοδολογία χρησιμοποίησαμε για τη μελέτη. Ε, desk review κυρίως, δηλαδή αναλύσαμε το ίμιση των προγραμμάτων που είχαν εγκριθεί μέχρι τότε δεν είναι μεγάλος ο χάρτης, αλλά το πράσινο είναι οι περιοχές που καλύψαμε με την ανάλυση μας. Ε, αναλύσαμε τα έγγραφα, τα παραστατικά των προγραμμάτων δηλαδή και για να ξέρουμε πώς, ποια είναι η αντίληψη των δικαιούχων και όσων ενεπλάκησαν στα προγράμματα. Ε, συζητήσαμε με ε, ε, τις διαχειριστικές αρχές και μέλη της γραμματείας. Για να περάσουμε τώρα στα βασικά πορίσματα ανά θέμα ε, τα αποτελέσματα και η σχετική προσέγγιση, τα ε, η στρατηγική συνοχή και ούτω καθεξής. Αρχίσουμε, θα πάρουμε τη σειρά. Στρατηγική συνοχή. Τα προγράμματα που παρουσιάσαμε σχετίζονται με μια στρατηγική που ε, προϋποθέτει συμμετοχή πολλών εμπλεκομένων φορέων. Ε, πολύ σημαντικό έβριμα της μελέτης μας. Όλες οι αναλυθήσεις στρατηγικές δείχνουν ισχυρή θεματική συγκέντρωση. Δηλαδή συνάδουν με το άρθρο 6 του κανονισμού ETC. Και είναι περιορισμένα ε, τα θεματικά πεδία και προτεραιότητες για τις επενδύσεις. Βλέπετε μια γενική επισκόπηση των θεματικών στόχων των προγραμμάτων που επιλέξαμε. Ε, ας πάρουμε το στόχο του περιβάλλοντος. Ε, έχουν ιδιαίτερη σημασία, ε, κυρίως ε, ο ρυθμός 6 ε, αλλά και 1 για την καινοτομία. Περισσότερα από τα μισά προγράμματα επέλεξαν αυτό το στόχο. Για να περάσουμε στο δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό της περίοδου 2014-2020 του ρυθμιστικού πλαισίου. Ε, βασιζόμαστε στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Αυτή είναι η προσέγγιση μας και λοιπόν σε αυτή την προγραμματική περίοδο ε, ζητούμε τεκμήρια για το αν ε, έχουν χρησιμοποιηθεί με καλή επιστροφή τα, τα, κονδύλια. Ποια σημασία έχουν για τη, τις περιοχές και επίσης ε, συστήματα εποπτείας παρακολούθησης ε, για να έχουμε ξαναλέω αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα ως προς τη χρήση των κονδυλίων μέσα στα προγράμματα. Αυτά σχετίζονται και με τα συγκεκριμένα προγράμματα αίτηση και με την ανάλυση μας. Καταδεικνύεται ότι τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας μπόρεσαν να, να συμμορφωθούν με αυτούς τους κανόνες. Με τα προγράμματα που αναλύσαμε αποδεικνύεται η προσπάθεια που γίνεται να βασιζόμαστε σε αριθμητικά, ποσοτικά, ποιοτικά, στατιστικά στοιχεία, σε αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και πρόγραμμα παρακολούθησης βάση των βασικών απαιτήσεων ε, του κανονισμού. Όμως, όμως και το τονίζουμε, οι ερωτηθέντες μας είπαν ότι υιοθέτησαν μια παρεμφερή προσέγγιση αλλά ήταν πολύ σημαντική πρόκληση για αυτούς. Γιατί, ακριβώς λόγω των χαρακτηριστικών της πολιτικής συνοχής, θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Για να έχουμε στρατηγικές που βασίζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες ε, των εδαφικών μονάδων, τι είναι σημαντικό. Τα ποσοτικά στοιχεία, στατιστικά στοιχεία. Οι ερωτηθέτες, λοιπόν μας υπέδειξαν ότι δεν είχαν ε, αρκετή, αρκετά δεδομένα σε επίπεδο νατς 3 κυρίως, ε, γιατί, κυρίως για τα διασυνοριακά προγράμματα και για τη συνεργασία με τρίτες χώρες τα στατιστικά δεδομένα ούτε καν ήταν διαθέσιμα. Σημαντική δυσκολία αντιμετώπισαν ως εκ τούτου και μπόρεσαν να συμμορφωθούν με τις απαιτήσει του κανονισμού, όμως χρειάζεται και να προσπαθήσουν πάρα πολύ και να δεχτούν βοήθεια από εξωτερικούς συμβούλους. Σε κάποιες περιπτώσεις ο δείκτης του 12-29 για το κοινό output, που πρέ, δείκτης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για, την εδαφική συνεργασία, τι γίνεται. Δείχνει πως δεν φαίνονται τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης που χρηματοδοτείται. Δεν πρόκειται για mainstream προγράμματα ε, σε εθνικό επιφερειακό επίπεδο. Μιλάμε για συγκεκριμένα προγράμματα εδαφική συνεργασία. συνέργειες. Όλα τα προγράμματα που αναλύσαμε δείχνουν ότι υπάρχουν πιθανές, ε, συνδυασμοί με άλλα όργανα με τον Ορίζοντα 2020, με το Κόσμε, με το Erasmus Συν. Αλλά αναφέρθηκαν και mainstream προγράμματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Περιορισμένος είναι ο αριθμός των προγραμμάτων που αναφέρεται σε άλλες στρατηγικές ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλα εργαλεία πέραν από τα εργαλεία της πολιτικής που σχετίζονται με τα ταμεία της Ένωσης. Σημαντικό είναι να τονίσουμε πως πέρα από την αναφορά στις πιθανές συνέργειες, ο τρόπος που στην πράξη ε, θα αναπτυχθούν τέτοιες συνέργειες ε, κατά τη διάρκεια ζωής του προγράμματος δεν ε, είναι προφανής, οπότε υπάρχουν όρια σε αυτά που μπορούν να επιτευχθούν. Απλούστευση. Το τωρινό αριθμιστικό πλαίσιο ε, περιέχει διάφορους τρόπους απλοποίησης για την ε, διοίκηση και για τους δικαιούχους. Τουλάχιστον αυτό είχε κατά νου ο νομοθέτης. Με την ανάλυση μας φαίνεται πως τουλάχιστον το 50% των προγραμμάτων περνώντας από τη μία προγραμματική περίοδο στην άλλη άλλαξαν τον τρόπο διαχείρισης χρησιμοποίησαν δυνατότητα όπως η συγχώνευση της διαχειριστικής αρχής και της αρχής πληρωμών. Και η σχέση ανάμεσα στη διοίκηση και τους δικαιούχους. Έχουμε αυτό το σύστημα ηλεκτρονικής συνοχής, ε, ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους δικαιούχους. Ε, υιοθετήθηκε από τα περισσότερα προγράμματα. Έκρινα πολύ χρήσιμο να έχουν στη διάθεσή τους το πρόγραμμα ε, το, ε, της Interact με τα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε προγράμματος βέβαια. οι, ε, τα SEOs, ε, απλουστευμένες αναλλακτικές λύσεις για το κόστος, θεωρούνται ως βασική λύση για τη μείωση του διοικητικού κόστους ε, και άχθους για τη διοίκηση και για τους δικαιούχους. Σε αυτό το στάδιο βλέπουμε ότι πολλά προγράμματα έχουν προκρίνει αυτά τα SEOs. Νέα εργαλεία εφαρμογής. Ε, CLLD, ε, δαφικές επενδύσεις, κοινό πρόγραμμα δράσης, ε, χρηματοοικονομικά εργαλεία, όλα αυτά είναι στη διάθεση των δικαιούχων. Όμως πολύ λίγα προγράμματα τα χρησιμοποίησαν τελικά αυτά τα εργαλεία. Γιατί έκαναν αυτή την επιλογή. Διότι θεωρούν, εκλαμβάνουν ως υπερβολικά ε, περίπλοκα αυτά τα εργαλεία να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της εδαφικής συνεργασίας. Μας είπανε οι ερωτηθέντες πως αυτά τα εργαλεία είναι καλά για τα mainstream προγράμματα, όχι για την, τα ETC, τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας. Συστάσεις. Μετά από αυτά τα απορίσματα θα συνοψίσω κάποιες ε, συστάσεις, ε, κάποιες για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, κάποιες ε, εστιάζονται περισσότερο στην περίοδο πέραν του 2020. Επειδή κάποια θέματα έχουν ιδιαίτερη σημασία, απλοποίηση και κυρίως αυτές οι νέες απλοποιημένες εναλλακτικές για το κόστος, φαίνεται να έχουμε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Προσπαθούμε να τονώσουμε την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών για τη χρήση αυτών των ε, options. Γιατί φαίνεται, όπως σας είπα, να είναι η λύση κλειδί που απλοποιεί τη ζωή όλων και τη διοίκηση και των δικαιούχων. Πέρα από τα SEOs, έχουμε τις κρατικές προμήθειες, ε, τις κρατικές επιδοτήσεις και τις νέες κατευθυντηρίες γραμμές και αυτές ήταν πολύ χρήσιμες. Δεν ξέρουμε όμως, όπως σας είπα, στην πράξη πώς θα υλοποιηθούν συνέργειες με άλλα εργαλεία. Χρειάζονται λοιπόν κατευθυντήριες γραμμές. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν ε, συνέργειες με άλλα μέσα. Μετά. Για τον προσανατολισμό, στατικό προσανατολισμό. Ε, κοιτάξαμε διαπιστώσαμε ε, τα επίπεδα στα οποία συμμετείχαν οι τοπικοί εμπλεκόμενοι φορείς ε, κατά το σχεδιασμό αλλά και κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων αλλά αποτιμήσαμε και την ικανότητα των προγραμμάτων να εποφεληθούν από τις διατάξεις απλοποίησης αυτές είναι οι συστάσεις για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, για την μελλοντική. Επανερχόμαστε σε κάποια ζητήματα σε σχέση με τον προσανατολισμό επί των αποτελεσμάτων. Κάποια προγράμματα ETC δυσκολεύουν να συγκροτήσουν μηχανισμούς παρακολούθησης. Ενδεχομένω θα μπορούσε να ενταθεί η προσπάθεια να βελτιωθεί ο δείκτης ε, κοινού αποτελέσματος, common output, ούτως ώστε να υπάρξει πιο ομοιόμορφη εφαρμογή στο τομέα της εδαφικής συνεργασίας. Ε, επίσης, θα πρέπει να καλύψουμε το χάσμα των στατιστικών δεδομένων, να συλλέξουμε στατιστικά στοιχεία εκεί που δεν υπάρχουν. Τελική σύσταση. Λόγω των δυσκολιών για τα νέα εργαλεία υλοποίησης, προτείνουμε να παραμείνει προαιρετική η χρήση τους. Αυτά είναι τα βασικά πορίσματα και οι συστάσεις. Είμαστε στη διάθεσή σας. Αν έχετε ερωτήσεις, θέλετε διευκρινήσεις, ε, οτιδήποτε. Εδώ είμαστε εμείς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ε, έχουμε ολοκληρώσει με την παρουσίαση. Ωραία. Συνάδελφοι ερωτήσεις, παρατηρήσεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για αυτήν την ε, εξαιρετική παρουσίαση. Ε, αυτό που εγώ συγκράτησα είναι ότι έχουμε επαναλαμβανόμενα προβλήματα. Όλοι μας διαμαρτύρονται σχετικά με την ε, απλούστευση και την απορρόφηση. Οπότε σας ρωτώ, έχετε εντοπίσει συγκεκριμένα αυτά βήματα, μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν στη συζήτηση αυτή, γιατί η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των διαφόρων δομών θα μπορούσε να είναι μία από τις λύσεις, αλλά εσείς έχετε εντοπίσει ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζονται προς την κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις. Παρακαλώ κύριε Ρόπε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να σχολιάσω ένα-δύο πράγματα, γιατί εδώ και αρκετά χρόνια έχω συμμετάσχει στην απορρόφηση και χρησιμοποίηση των ε, διαφορετικών ταμείων και ταμείων συνοχής. Και ακούω ξανά και ξανά τα τελευταία χρόνια τον όρο απλούστευση. Το είχα ακούσει στην προηγούμενη εντολή, στη χώρα μου, το ακούω και τώρα αυτό που βρίσκω ενδιαφέρον είναι και θα ήθελα και την άποψη της Κομισιόν σχετικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα όταν υλοποιηθεί αυτή η δουλειά. Όταν μιλούμε για την περίοδο 14-20 πρέπει να θυμόμαστε ότι στην υφιστάμενη περίοδο τα προγράμματα, τα έργα δεν έχουν υλοποιηθεί. Είμαστε στη φάση της όρευσης προτάσεων, ιδεών και εγγράφων. Τουλάχιστον στη Λιθουανία από την οποία και προέρχομαι οι διαγωνισμοί θα ξεκινήσουν μόλις του χρόνου και αυτό είναι το πιο αισιόδοξο σενάριο. Και η οποιαδήποτε απορρόφηση θα ξεκινήσει, εάν ξεκινήσει, μόνο στο δεύτερο ήμιση της περίοδου 14-20. Αυτό θα το δούμε κάποια στιγμή ή δεν έχουμε σκοπό Γιατί λέμε 2 συν 3 δεν θα έπρεπε να προετοιμαζόμαστε ήδη για τη νέα περίοδο. Για να μπορούμε όταν ξεκινάει η περίοδος, εκ των προτέρων εννοώ, ώστε να μπορούμε όταν ξεκινάει η περίοδος να χρησιμοποιούμε τα ταμεία. Ιδάλλως πρέπει να χρησιμοποιούμε τα προηγούμενα κονδύλια για δύο ή τρία χρόνια. Η ροή, η εισρωή ροή ειναι τεράστια οι τιμές αυξάνονται στο μεταξύ και δημιουργούνται κενά. Δεν υπάρχει χρόνος πλέον να υλοποιηθεί το πρόγραμμα και υπάρχουν και μεγάλα κενά αδράνεια όπου δεν υπάρχουν πόροι οι διάφοροι φορείς, διαχειριστές, αναλυτές κτλ. τα λοιπά δεν έχουν πλέον δουλειά ενώ σε ορισμένα διαστήματα έχουν τόση πολλή δουλειά που δεν μπορούν να αντιχειριστούν σε άλλα διαστήματα δεν έχουν καθόλου. Δεν έχει καθόλου ομαλά το όλο πράγμα. και καλή η απλούστευση. Αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι τελικώς. Έχουμε λιγότερα σφάλματα. Έχουμε λιγότερα λάθη. Η περίοδος υλοποίησης έχει συντομευθεί. Σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε λιγότερους ανθρώπινους πόρους, ότι έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία, και στα κράτη-μέλη και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Γιατί ε, έχουμε 5 με 6 αρχές που διαχειρίζονται το κάθε ταμείο. Πέραν αυτών υπάρχει η κάθε μία από αυτές έχει τους δικούς της κανόνες, το κάθε ταμείο Δηλαδή χρησιμοποιείς ας πούμε πόρους για να προχωρήσεις σε μια επισκευή ενός κτηρίου από δύο διαφορετικά ταμεία για το ίδιο έργο, αλλά οι κανόνες είναι διαφορετικοί για τα δύο σετ κονδυλίων. Επομένως, μέσω της απλούστευσης θα έπρεπε να ενοποιήσουμε την αιρεσιμότητα της προϋποθέσης. Γιατί κάποια ταμεία προκαταβάλουν κονδύλια, άλλα ταμεία μόνο αποσημειώνουν για καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κτλ. Και οι άνθρωποι που εργάζονται στο πεδίο, που ασχολούνται με αυτά συνεχώς, δεν κατανοούν, δεν καταλαβαίνουν. Γιατί για την ίδια δουλειά έχεις διαφορετικές προϋποθέσεις. Και ο λόγος είναι ότι προέρχονται από διαφορετικά ταμεία. Και η εντύπωση, η μου είναι ότι αυτό έχει γίνει συνειδητά και σκοπίμως. Γιατί με περισσότερες προϋποθέσεις, όλο και περισσότερες προϋποθέσεις, ε, θα τολεπλασιάζονται και τα σφάλματα και τα λάθη και οι παραλήψεις. Ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψή σας σχετικά με όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάποιες άλλες επιθυμίες, παρεμβάσεις Κυρία Μαλέτσης, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση και για τα όσα ετοιμάστηκαν. Όταν κάνουμε λόγο για την περιφερειακή συνεργασία, καλό είναι να την αντιμετωπίζουμε την περιφερειακή συνεργασία και υπό το πρίσμα των ε, χρηστών και των εποφελούμενων. Είναι πολύ περίπλοκο διότι έχουμε κράτη-μέλη και μη κράτη-μέλη, έχουμε και διαφορετικούς κανόνες που ισχύουν σε σχέση με τα διαφορετικά προγράμματα. Υποβάλλουν αίτηση για ένα πρόγραμμα, μαθαίνουν κάποια πράγματα, υποβάλλουν αίτηση για άλλο πρόγραμμα, πρέπει να μάθουν καινούρια πράγματα και υπάρχει σύγχυση που δημιουργείται και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κάποιο μεγάλο όφελος τώρα όταν προσθέτουμε αυτό το νέο μέσο για την ε, υλοποίηση το οποίο αναλύθηκε, βλέπουμε ότι είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να υπάρχει σωστή εφαρμογή και υλοποίηση από τα κράτη-μέλη, διότι έχουμε διαφορετικούς κανόνες, διαφορετικά προγράμματα. Διαρωτώ με, σε σχέση με αυτή την ανάλυση, πώς καταλήγουμε σε πιθανά συμπεράσματα ότι γίνεται η προσπάθεια να υπάρξει μικρότερη παραλλαγή σε σχέση με τα περιφερειακά προγράμματα, σε σχέση με τους κανονισμούς μας και πώς μπορούν να πλουστευθούν περισσότερο. Η σύστασή σας είναι σαφής. Χρειάζονται νέες κατευθυντήριες γραμμές, new guidelines, για να μπορέσουν όλα αυτά τα καινοτόμα στοιχεία τα οποία από το 2014 έως το 2020 θα εισαχθούν και θα λειτουργήσουν όταν αρχίζουν όμως νέες τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές, εκατοντάδες σελίδες υποβάλλονται για το πώς θα πρέπει να λειτουργήσουν όλα αυτά και είναι πραγματικά δύσκολο να τα μάθουν οι χρήστες όλα αυτά. Πρέπει να απλουστευτούν αυτά πρόκειται για, τον, για θέματα προϋπολογισμού και πρέπει να διασφαλιστούν κάποιες δράσεις προτού ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα. Και τώρα να εξοικειωθεί κανείς με όλα αυτά πώς είναι δυνατόν με τόσα πολλά καινούργια πράγματα και τόσες νέες καινούργιες διατάξεις να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Ευχαριστώ. Κύριος Φανίστερ Ρόι, σας ευχαριστώ για αυτές τις πληροφορίες. Μια πιο γενικού χαρακτήρα ερώτηση θα είχα, Πρόεδρε, που θέλω να διατυπώσω. Στην Ολομέλεια μόλις συγκρίναμε την έκθεσή σας και τώρα έχουμε και την μελέτη και πολλές ε, ουσιώδεις ε, παρατηρήσεις ε, που σε σχέση με το σχεδιασμό και την έκβαση μελετών δεν θα έπρεπε να περιμέναμε ίσως δύο-τρεις μήνες καλύτερα να δούμε τι θα έπρεπε να γίνει δεν είναι μόνο το θέμα του να υπάρξει κάποια δραστηριοποίηση απλά και μόνο χάρη της απασχόλησης κάποιων. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Φυσικά θα τοποθετηθώ σε αυτό που είπατε. Επιτρέψτε μου στο τέλος λοιπόν και εμένα να πω σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συμμεριστώ σε σχέση με τον κύριο Φανίστερ και τους συναδέφους στις δικές μου σκέψεις. Ναι, νομίζω ότι θα μπορούσαν τα πράγματα να είχαν οργανωθεί καλύτερα. Θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη προτού ξεκινήσαμε την έκθεση ε, ιδίας πρωτοβουλίας. Αλλά επίσης και μια μελέτη της Επιτροπής θα μπορούσαμε να είχαμε πριν από τη δική μας έκθεση. Όπως θα θυμόσαστε, είχαμε μία καθυστέρηση πρόταση στη συζήτηση για την έκθεση επειδή αναμέναμε τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Συνεργασία και ποτέ δεν ε, κατατέθηκε, δεν δόθηκε αυτή η μελέτη. Και τώρα βλέπουμε αυτή τη μελέτη. Πολύ καλό αυτό. Χαίρομαι πολύ για το ότι υπάρχει μια τέτοια μελέτη για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Συνεργασία, European Territorial Cooperation. Τα περισσότερα θέματα τα οποία συζητήσαμε στην έκθεσή μας εδώ στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης τα βλέπουμε να αναφέρονται τώρα στη μελέτη αυτή. Δυστυχώς όμως κάποια από αυτά με κάποιο αρνητικό πρόσημο η τάση. Επειδή εγώ στη δική μου έκθεση με μεγάλη προσοχή που επένδυσα για αυτό το νέο μέσο, το νέο εργαλείο για τη συνέργεια, για το χρηματοοικονομικό μέσο, για όλα αυτά τα νέα μέσα και εργαλεία φιλόδοξα. Τώρα λέτε ότι ένας πολύ περιορισμένος αριθμός των προγραμμάτων κάνουν χρήση αυτού του μέσου και δεν σχεδιάζουν να κάνουν χρήση και στο μέλλον ακόμα αυτού του μέσου. Φαίνεται ότι τα διαμεθοριακά προγράμματα είναι ιδιαίτερα περίπλοκα επειδή έχουν και διαφορετικό χαρακτήρα. Έχουμε περιφέρειες στη Βουλγαρία που σε σχέση με αυτό το ένα πρόγραμμα για παράδειγμα μεταξύ δύο κρατών και έχουμε και το πρόγραμμα με τη Μακεδονία για παράδειγμα και άλλα παραδείγματα από άλλες ε, περιοχές της χώρας. Αυτά τα προγράμματα είναι τελείως διαφορετικά λοιπόν μεταξύ τους και η διαχείρισή τους είναι πολύ διαφορετική. Πώς να γίνει λόγος λοιπόν για απλούστευση, πώς να γίνει λόγος για τα νέα εργαλεία και μέσα και για τη συνέργεια και πώς μπορεί να γίνει λόγος για πολύ πιο φιλόδοξους στόχους ε, και διαδικασίες για να χρησιμοποιηθεί αυτό το νέο μέσο της, ε, που θα χρησιμοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων για παράδειγμα προς όφελος αυτών των δράσεων. Απόλυτα λοιπόν συμφωνώ μαζί σας ότι είναι ένα ζήτημα ετοιμότητας των κοινοτήτων και των όσων θα επωφεληθούν από όλα αυτά. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε να προετοιμαστούν μόνοι τους όσοι θα επωφεληθούν από αυτά τα προγράμματα. Πρέπει να επενδύσουμε στην περιφερειακή συνεργασία. Και αυτό επειδή αυτή είναι μία από τις κατευθύνσεις που πιστεύω ότι μπορούμε έτσι να αναπτύξουμε την περιφερειακή πολιτική στο μέλλον πρέπει να επενδύσουμε και στην τεχνική αρρωγή. Είδα κάποια στοιχεία από πλευρά των εγγράφων. Είναι τόσο περιορισμένη αυτή η τεχνική αρρωγή, η τεχνικού χαρακτήρα αρρωγή για κάποια από αυτά τα προγράμματα, απίστευτα περιορισμένη. Και λαμβάνοντα υπόψη τα, τις παρεμβάσεις και τις ερωτήσεις των συναδέλφων, είναι τεράστια σπουδαιότητα να αντιληφθούμε ότι πρέπει αυτή η τεχνική αρρωγή να αυξηθεί οπωσδήποτε. Σε κάποια σημεία συνδέεται αυτό με την προηγούμενη συζήτηση επίσης. Με την προηγούμενη συζήτηση και αυτό διότι ε, γίνεται λόγος για διαθροτικές μεταρρυθμίσεις. Γίνεται λόγος για μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη και σε, στις διαμεθοριακές περιοχές και χρειάζεται η συνδρομή και η υποστήριξη της τεχνικής αρρωγής. Αν δούμε τους κανόνες και κανονισμούς για αυτή την τεχνική αρρωγή <clears throat> πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε μια μεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε στο μέλλον και σε συνδυασμό με την προηγούμενη συζήτηση για την υποστήριξη από τα διαθροτικά ταμεία με το προηγούμενο πρόγραμμα. Συγγνώμη, μακρηγόρησα ίσως, αλλά αφορά την έκθεσή μου αυτό το θέμα. Αν θέλετε να αντιδράσετε, παρακαλώ έχετε τον λόγο. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω την εντύπωση ότι τα τρία ερωτήματα έχουν ένα συσχετισμό. Πώς απλουστεύουμε, πώς αναρμονίζουμε καλύτερα ώστε να διευκολύνουμε τους δικαιούχους. Αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω λοιπόν εδώ είναι τα δεδομένα που έχουμε αναλύσει αλλά και την εντύπωση που αποκομίσαμε από τους ερωτηθέντες, διαχειριστικές αρχές, γραμματείες κτλ όπου έχουν σημαντική εμπειρία στη διαχείριση των προγραμμάτων αυτών. Αυτό που μπορώ να σας πω λοιπόν για την εναρμόνιση. Το γεγονός ότι οι δικαιούχοι πολύ συχνά έχουν να αντιμετωπίσουν τελείως διαφορετικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα μία. Εδώ εγώ βέβαια μπορώ να εστιαστώ μόνο στα πλαίσια της εδαφικής συνεργασίας. Αλλά έχω την εντύπωση ότι σε αυτήν τη νέα προγραμματική περίοδο καταβάλουμε, καταβάλλεται με αλφαγιώτα μία προσπάθεια του να είμαστε όσο πιο εναρμονισμένοι μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων γίνεται. Η παραπομπή στα συστήματα ελέγχου και επιτήρησης είναι ένα καλό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας κοινή προσέγγισης στην επικοινωνία με τους δικαιούχους. Η απλούστευση τώρα που είναι ένα τεράστιο ζήτημα και πάλι η εντύπωση που έχω από τα πορίσματα είναι ότι υπάρχει ευρύτερη συνένεση ότι παρακτική λύση που ήδη είναι διαθέσιμη παρέχεται από το άρθρο 67 του CPR και το 19 και είναι η χρήση του επιλεγμένου κόστους του απλουστευμένου, με συγχωρείτε, της επιλογής του απλουστευμένου κόστους. Αυτό διευκολύνει σημαντικά τον δικαιούχο και εξασφαλίζει και λιγότερη πιθανότητα σφαλμάτων. Είναι ένα σαφέστατο πόρισμα προκύπτει από τη μελέτη. Και είναι πολύ σημαντικό σημείο κίνηση. Δηλαδή, οτιδήποτε μπορεί να γίνει προκειμένου να διευκολύνει την επιλογή του οπισθωμένου κόστους απλουστεύει και διευκολύνει τα πράγματα. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Φρανσουά, ο οποίος θα συνεχίσει στα γαλλικά. Κοιτάξτε, δεν πάνε όλα άσχημα. Οι διαχειριστικές αρχές ε, που ρωτήσαμε λένε ότι η συγκέντρωση επί κάποιων θεματικών των ταμείων λειτουργεί αρκετά καλά. Έχει γίνει κατανοητό από τους εταίρους, από τους χρήστες, Από εκεί πέρα όταν πρέπει να επιτηρήσει κανείς να παρακολουθήσει τα προγράμματα, Πράγματι, έχουμε περίπλοκους ε, δείκτες, καμιά φορά δεν έχουμε τους κατάλληλους ίσως δείκτες, αλλά επί του θέματος της συγκέντρωσης, λέει ο δεν είχαμε αρνητικά σχόλια και παρατηρήσεις, αντίθετα. Έχουμε προβλήματα επί των νέων μέσων, ναι, αλλά εδώ είμαστε σε ένα πλαίσιο διασυνοριακής και διακριτικής συνεργασίας που είναι ήδη, έχει τις ιδιαιτερότητές του είναι διάφοροι φορείς που παρεμβαίνουν στη συζήτηση και στον πραγματισμό Γιατί βεβαίως η μελέτη μας επικεντρώθηκε στον προγραμματισμό. Έχουμε λοιπόν διάφορα επίπεδα εκεί παρέμβασης. Ήδη το μέσο ε, ε, είναι ε, σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένο. Δηλαδή συμπεριλαμβάνει πάρα πολλούς φορείς και αρμοδίους. Και επομένως ε, ε, οι προσεγγίσεις της, ε, του ολοκληρωμένου προγραμματισμού είναι ενδεχομένως λίγο πιο δύσκολες στην κατανόησή τους. Πάντως η, η εντύπωσή μας είναι, γιατί όπως είπε και ο συνάδελφος δίνουμε μια εικόνα, είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα βαθμό περιπλοκότητας που καλό θα ήταν να μην τον ξεπεράσουμε. Εγώ θα ήμουν υπέρ των guidance Καλό θα ήταν δηλαδή στις διαχειρικές αρχές να παρέχουμε ε, ε, εκείνα τα εργαλεία που χρειάζονται χωρίς βεβαίως να αλλάζουμε τελείως τον κανονισμό. Δηλαδή να δίνουμε στους υπευθύνου τα μέσα εκείνα που θα τους χρειαστούν για να διαχειριστούν το πρόγραμμα. Γιατί σε τη φάση της αξιολόγησης πρέπει να αξιολογήσουμε και πολύ προσεκτικά το τι έχει συμβεί και πράγματι για τις συνέργειες μεταξύ των διαφορών μέσων, ναι, έχουμε πολλά μέσα. Πολλές διευκολύνσεις, πολλά ταμεία και καμιά φορά είναι δύσκολο για τον δικαιούχο που υποβάλλει το πρόγραμμά του. Υπάρχουν διάφορες κλίμακες, ε, πίνακες, ε, κανόνες κτλ. που πολύ συχνά είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς γιατί αλληλεπικαλύπτονται. Δεν υπάρχει σε κάθε περίπτωση μαγική λύση, γιατί δεν είμαστε στην εκκίνηση των προγραμμάτων μεν, αλλά ούτε έχουμε φτάσει στην πλήρη υλοποίησή τους ώστε να έχουμε ενδείξει αποτελεσμάτων. Αυτά θα είχα εγώ να πω από πλευρά μου. Σα ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Να έχετε κάτι ακόμα ή να θεωρήσω Έχουμε κάποιον από την Κομισιόν που θα ήθελε το λόγο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω για αυτήν πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που έρχεται στη, στην κατάλληλη χρονική στιγμή γιατί προετοιμαζόμαστε για την μελλοντική εξέταση. Θα ήθελα να πω ότι μας ανησυχούν τα ζητήματα που, που η έκθεση υπογραμμίζει ε, η καθυστερημένη απορρόφηση επίσης πολλών από τα προγράμματα και ενθαρρύνουμε τις διαχειριστικές αρχές να ξεκινήσουν να προχωρήσουν στην πραγματική υλοποίηση. Κατανοούμε ότι καθότι η διαδικασία της ανάθεσης δεν έχει ολοκληρωθεί σε πολλές από τις περιπτώσεις ε, θα συνιστούσαμε στα κράτη-μέλη να ολοκληρώσουν η διαδικασία των αναθέσεων. Τώρα, εμείς είμαστε οπωσδήποτε υπέρ της μεθόδου του απλουστευμένου κόστους. Αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν το έχουν υιοθετήσει όλες οι διαχειριστικές αρχές. Άρα λοιπόν η πρόταση κομισιών στον κανονισμό Omnibus έχει, ενέχει και άλλες κατευθύνσεις χρήσεως για το αποσταγμένο κόστος ώστε να το καταστήσει υποχρεωτικό για προγράμματα που λαμβάνουν κάτω των 100.000 ευρώ. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό για πάρα πολλά μικρής κλίμακας έργα και που θα έχει αντίκτυπο για την εναρμονισμένη χρήση των ε, μέσων υλοποίησης βλέπουμε και εδώ τη θετική εξέλιξη ότι όλο και περισσότερα έργα χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Υπάρχει δηλαδή μια εναρμόνιση και αυτό βοηθάει τους δικαιούχους. Για τις δε βελτιωμένες συνέργειες ε, ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να υλοποιούν εκείνες τις δράσεις που προβλέπονται καθότι όλα υποχρεούνται να περιγράφουν για τους μηχανισμούς υλοποίησης πώς εξασφαλίζονται οι συνεργασίες με τα μέσα κοινωνικής, ε, ε ναι, πολιτικής κοινωνικής συνοχής και άλλα που χρησιμοποιούν. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Now I can Ευχαριστούμε. Ολοκληρώνουμε έτσι τώρα τις συζητήσεις. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και την Επιτροπή για την συμμετοχή της. Ευχαριστώ συνάδελφοι για τη συζήτηση. Ήταν το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξή μας. Το επόμενο είναι η έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών. Λάβατε τις αποφάσεις τους. Υπάρχουν αντιρρήσεις, ενστάσεις στο σχέδιο, στα συμπεράσματά τους. Όχι. Εγκρίνονται λοιπόν οι αποφάσεις των συντονιστών. Τώρα διάφορα. Υπό τα διάφορα υπάρχει κάτι. Δεν παρίστασε ο κύριος Φανίστερ Ρόι, οπότε δεν έχουμε και διάφορα θα έλεγα. Δεν έχουμε λοιπόν άλλα. Και να υπενθυμίσω τις επόμενες συνεδριάσεις. Αύριο θα έχουμε την κοινή συνεδρίαση το απόγευμα 2.30 στην, στο κτίριο της Επιτροπής Περιφερειών. Η επόμενη συνάντηση Τετάρτη 9η Νοεμβρίου από τις 3 ε, το απόγευμα και πέμπτη <clears throat> επόμενη ε, συνεδρίασή μας ε, στις 9 το πρωί. Αυτά από πλευράς μου ως ενημέρωση. Ευχαριστώ τους διερμηνείς για τη βοήθειά τους στο έργο μας σήμερα. Σας ευχαριστώ. Λίγη συνεδρίαση της Επιτροπής μας για σήμερα. Γεια σας.